17 Απριλίου από τις 9 το πρωί και μετά στις 3 το απόγευμα. Η μέση διαταξή έχει δημοσιευτεί στο διαδίκτυο και τα πρακτικά επίσης θα δημοσιευτούν. Ευχαριστώ. Καληνύχτα.